για μια σύντομη ανακοίνωση την οποία θέλω να κάνω. Meine Damen und Herren, in diesen Minuten... Αυτές τις στιγμές, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Αλγερία έχει οξυνθεί δραματικά. Ο Αλιενός στρατός έχει αντιμετωπίσει να αντιμετωπίσει την Αΐνα Μενάσα, η οποία είναι μια ένοπλη ομάδα, η οποία έχει συλλάβει Ευρωπαίους ε, ε ομήρους. Η κατάσταση λοιπόν γίνεται ε, όλο και πιο οξία. Έχει σκοτωθεί ένας Βρετανός όμηρος και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε εμείς στην οικογένειά του και στη Βρετανική κυβέρνηση να εκφράσουμε την ε, συμπαράστασή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταξύ των ομήρων ε, Αλγερινούς αλλά και Ευρωπαίους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας μαζί τους και ελπίζουμε ότι οι Αλγερινές αρχές θα κάνουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να απελευθερθούν το ταχύτερο δυνατό. Αυτή η κατάσταση δείχνει πόσο έντονες είναι οι αντιπαραθέσεις στο Σαχέλ. Υπάρχει η απειλή των τζιχαδιστών η οποία συνεχίζεται. Δεν πρόκειται μονάχα για μια απειλή για αυτή την περιοχή, αλλά είναι μια απειλή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και για την ειρήνη στο σύνολο της περιοχής της Μεσογείου. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω ότι θα υπάρξει ειρηνική απόλυξη αυτής της ομοιρίας χωρίς περαιτέρω θύματα. Κυρίε και κύριοι, η διαδικασία του άρθρου 70